Επόμενο σημείο έχουμε των ε, μέτρων για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ Καταρχήν οι συντάκτες του ψηφίσματος ξεκινάμε με τον κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα για 1,5 λεπτό. Όλα τα ανθρώπινα όντα γεννούνται ίσα με την ίδια αξιοπρέπεια και τα ίδια δικαιώματα και έχουν την υποχρέωση να μην προωθήσουν τη βία επί τη βάση ατομικών χαρακτηριστικών όπως είναι η σεξουαλική έκφραση και το φύλλο. Είναι απαραίτητο λοιπόν όλες οι χώρες να εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να μην ποινικοποιούν τις ε, σεξουαλικές δραστηριότητες μεταξύ συνενούντων ε, ενηλίκων. Σε πολλές χώρες υπάρχει κολασμός των ομοφιλοφιλικών δρασέων μεταξύ ηλικιωμένο σε χώρες όπως η Ουγγάντα και σε χώρες όπως η Νιγηρία. Γι' αυτό στο ψήφισμα αυτό εμείς θέλουμε να καταδικάσουμε το γεγονός ότι εγκρίνονται όλο και περισσότεροι καταπιεστικοί νόμοι κατά των ΛΟΑΔΜ και τονίσουμε ότι η σεξουαλική ταυτότητα είναι, θέματα, είναι ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο. Ζητούμε λοιπόν από όλες αυτές τις χώρες να σταματήσουν την ποινικοποίηση των ε, σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και να ζητούμε από τον πρόεδρο της Ουγγάντα να μην εγκρίνει την υπογραφή αυτού του νόμου και το ίδιο πράγμα στην Ιγυρία. Ζητούμε επίσης από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να έχουν μια εκπεφεσμένη ρήτρα για την μη ε, αποδοχή της ποινικοποίηση αυτής στα, στην επόμενη αναθεώρηση της Συμφωνίας, Συμφωνίας Κοτονού, όπως το έχουμε πράξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέδα και Ρουέδα. Ακολουθεί ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων όσο προχωρούν στην Ευρώπη φαίνεται ότι υποχωρούν σε άλλες χώρες του κόσμου. Βλέπουμε ότι σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου υπάρχουν ε, διακριτικές μεταχειρήσεις των ΛΟΑΔΜ. Στην Ινδία ας πούμε αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχουν απικιακής εποχής και τύπου νομοθετήματα τα οποία τα ξαναθυμούνται και τα ξαναφέρνουν στην επιφάνεια. Ε, τα δικαιώματα βεβαίως έχουν την δυνατότητα χωρίς καμία εξωτερική ε, ανάμιξη να ε, κάνουν τα νομοθετήματά τους. Απλώς θα πρέπει να προβλέπονται και εναλλακτικέ μορφές για τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Νομίζω ότι θα πρέπει πρέπει να ε, συνεργαστούμε με όλους τους φορείς αυτών των χωρών, αναφέρομαι κυρίως δε στην Ουγκάντα και την Νιγηρία, έτσι ώστε να σταματήσει η προώθηση αυτών των ε, κακών και δυσάρεστων νόμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Ακολουθεί κυρία Σάκη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπα, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάρα πολλές προκλήσεις αντιμετωπίζουν η κατηγορία των ατόμων ΛΟΑΔΜΟ εξαιτία νόμων που τους καταδικάζουν, καταδικάζουν την ταυτότητά τους, περιορίζουν δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και αυτό είναι ακόμα πιο ενοχλητικό, επειδή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να είναι δύσκολο να πετύχουμε να καταδικάσουμε όλοι μαζί τις παραβιάσεις που γίνονται σε βάρος τους. Είναι τροπή για την Ευρώπη σήμερα. Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνούνται να καταδικάσουν την Ρωσία για τα όσα κάνει σε βάρος τους είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό. Κυρίως μάλιστα τώρα που οι πολίτες μας βασίζουν τόσο πολλά σε εμά. Στη χώρα μου, στις κάτω χώρες για παράδειγμα, δείξανε το πραγματικό τους χρώμα όταν έστειλαν την ε, πιο σημαντική, το πιο σημαντικό κομμάτι των αθλητών να πάνε στην Ρωσία για να συμμετάσχουν εκεί στους χειμερινούς ε, Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να κάνουν το ίδιο μάλλον για τα άτομα αυτά και όχι για τους Ολυμπιακούς. Εγώ λυπούμε πολύ για το αποτέλεσμα αυτό. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι μας ατομικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αποτελούμε μέρος αυτών που προσπαθούν να πετύχουν την ισορροπία και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΟ. Είναι δικιά μας ευθύνη, γιατί τα δικαιώματα αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Για λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε 78 χώρες του κόσμου δεν αναγνωρίζονται ακόμα τα ε, δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και των λεσβιών. Ε, σε 7 χώρες ε, προβλέπεται ακόμα και η θανατική ποινή. Ωστόσο, στο Τσάντ, στην Μπουρκίνα Φάσο, στην Κεντρική Αφρική, στο Κονγκό, στην ε, ε, ε, Γουινέα, στην Μαδαγασκάρη, στο Μαλί, στην ακτή του Ελεφαντοστού, στη Ρουάντα και στην Νότια Αφρική. Έχει γίνει ήδη αποδεκτή η συνενετική πράξη μεταξύ ενηλίκων. Αυτό βεβαίως είναι αποτέλεσμα κοινών και μεγάλων προσταθειών. Στην Ουγγάντα, στην Ιγερία και με κάποιο άλλο τρόπο βέβαια η Ρωσία που δεν επιτρέπει πλέον ομοφιλοφιλική προπαγάνδα ε, ε, ε, οπισθοδρομούν. Έχουν υπογράψει νόμους που αποτελούν στην ουσία υποδάβληση του μίσους. Ζητούμε λοιπόν στις ενωσιακές αρχές να χρησιμοποιήσουν την μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση συγγνώμη, της Συμφωνίας του Κοτονού έτσι ώστε να εισαχθεί στη Συμφωνία αυτή η οποία να αναφέρεται σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα τόσο προσφυλή στην αριστερά που ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, απασχολήσουν ε, και όλο το πολιτικό τόξο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόουζα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Η Ινδία αλλάζει το σύνταγμά για να ποινικοποιήσει την ε, ομοφιλοφιλία. Η Ουγγάντα εγκρίνει ένα αντίστοιχο νόμο και η γερουσία της Νιγηρίας απαγορεύει την, ε, το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου, ακόμα και την ύπαρξη οργανώσεων ΛΟΑΔΟΜ. Στην Ρωσία, οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση υπέρ των ΛΟΑΔ είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, συνεχίζει την επίθεση κατά των ε, ομοφιλοφίλων. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από έντονες ενέργειες εναντίον των ΛΟΑΤΜ. Στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική δεξιά θέλει να ε, υπονομεύσει αυτό το δικαίωμα για τη σεξουαλική ταυτότητα. Θέλει να ε, κυνηγήσει τους ΛΟΑΔ. Υπάρχει όμως αυτή η βασική ε, ρήτρα ότι δεν πρέπει να αναμοχλεύουμε το, το μίσος εναντίον των των άλλων ανθρώπων. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μία νομοθεσία η οποία ε, θέτει τους ομοφιλόφιλους στη φυλακή αν δεν θέλουν ιατρική ε, υποτίθεται θεραπεία. Είναι απαραίτητο λοιπόν, απολύτως απαραίτητο να ξεπεράσουμε όλες τις προκαταλήψεις που έχουμε και να κατανοήσουμε την απλή ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο ζει κάποιος άλλος είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα α, ε, απαράδεκτο. Γιατί δεν μπορούν οι ΛΟΑΔΜΟΥ να έχουν οικογένειε με τη δική τους αντίληψη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή τη φοβία κατά των ΛΟΑΔΜ σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν δικαιώματα για όλους που είναι τα ίδια και είναι ίσα. Ευχαριστώ κυρία Σόουσα. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό ο κύριος Πρέδα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής διάκρισης που να βασίζεται στην εθνική προέλευση ή στην σεξουαλική προτίμηση. Πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά δεν υπέγραψα το κοινό ψήφισμα όσον αφορά το θέμα που συζητάμε τώρα. Και αυτό διότι πιστεύω ότι προσανατολίζεται περισσότερο στην προκλογική εκστρατεία και δεν έχει τόσο σχέση με τα κατεπήγοντα όπως συμβαίνει με άλλα θέματα που εξετάζουμε Εμάς μας απασχολεί περισσότερο ότι συμβαίνει στην Ουγκάντα, στην ε, Νιγηρία ή τη Ρωσία. Ζητάμε από τον πρόεδρο της Ουγκάντα να καταργήσει την παράγραφο 450 του ποινικού κώδικα της χώρας αυτής που θεωρεί έγκλημα την σεξουαλική αυτή το ίδιο και για το ποινικό κώδικα της Νιγηρίας. Τα άρθρα εκείνα δηλαδή, τα οποία αναφέρονται σε σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου. Η Ινδική κυβέρνηση ζήτησε όμως από το Δικαστήριο να αναθεωρήσει την απόφασή του σχετικά με την παράγραφο 377 του Δικού Ποινικού Κώδικα που απαγορεύει την ομοφιλοφιλία. Τέλος, όσον αφορά τη Ρωσία, καλά, σταματάω εδώ. Λέω ο μιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Αυτά για τους συντάκτες των ψηφισμάτων. Ερχόμαστε τώρα στις πολιτικές ομάδες. Με πρώτο τον κύριο Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα την Ευρώπη δεν ε, καταδικάζεται κανείς και δεν υφίσταται διακριτική μεταχείριση ε, για τις ε, σεξουαλικές του επιλογές. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις αρχές αυτές και στον υπόλοιπο κόσμο. Κυρίως στην Ουγγάντα και στην Νιγηρία ξέρουμε ότι η ΛΟΑΔΜ ε, αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Ε, νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα μέσω και της βοήθειας που δίνουμε στις ε, χώρες αυτές να ασκήσουμε πίεση Τώρα, μέσα στην Ευρώπη έχουμε και τη Ρωσία, η οποία είναι η βόρεια υπερδύναμη. Ε, αλλά όσο φαίνεται μεγαλώνει η δύναμη της, τόσο μικραίνει το μυαλό της και στενεύουν ε, οι απόψεις της. Ε, οπωσδήποτε αυτά αυτό που προσπαθούν να κάνουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς είναι απίστευτο και νομίζω ότι θα αποτελέσει κοιλίδα για όλους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μια τέτοια στάση. Πρέπει να την καταδικάσουμε όλοι. Για ένα λεπτό, Για ένα κυρία Γκόμε. Η ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ στη Λιγυρία, την Ουγγάντα, τη Ρωσία και την Ινδία που οδηγεί σε, φυλα... σε ποινές είναι μια σοβαρή απειλή στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να αναπτύξει κανείς την προσωπικότητά του. Είναι μια α, διάκριση κατά των ΛΟΑΔΜ και πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε αυτά τα άτομα τα οποία την χάνουν σοβαρών διακρίσεων σε διάφορα επίπεδα σε αυτές τις χώρες και σε άλλες και να συνεχίσουμε τον αγώνα για να διατηρήσουν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα διμερή και πολυμερή ε, φόρα που έχει για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ε, κινήσεις και να εξασφαλίσει ότι θα επηρεαστούν οι διμερείς σχέσεις με τις αμπλεκόμενες χώρες. Όταν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι οι οποίοι ε, εγκρίνονται σε χώρες που είναι εταίροι προνομιακοί μας με τη Συμφωνία της Κοτονού, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει κάποια μέτρα. Ζητούμε από την Κομισιόν να ξεκινήσει τη, δυνα... τη διαδικασία μεταρρύθμισης της συνδίκης της Κοτονού, λαμβάνοντας υπόψη τις διεκδικήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Για ένα λεπτό κύριος Μπένιον. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση, το ψήφισμα αυτό, γιατί είναι ανησυχητική η διάσταση που παίρνει η διακριτική μεταχείριση των ΛΟΑΔΜ. Ε, εφτά χώρες ε, προβλέπουν ε, την μέγιστη ποινή, θανατική καταδίκη για τους συνενούντες ενήλικες μεταξύ ατόμων του ιδίου ε, φύλου. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όντω η Συμφωνία Κοτονού ε, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτή η Συμφωνία ε, ε, έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να εκριζώσει την ένδια στην Αφρική. Ε, δεν θα πρέπει επομένως να καταργηθεί η συνθήκη αυτή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο πίεσης, αλλά κυρίως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και σαν τρόπος οικοδόμησης ικανοτήτων. Στο Birmingham, ας πούμε, έχουμε μια τέτοια προσπάθεια που έχουν αναλάβει ε, οι ε, ενώσει των ΛΟΑΔΜΟ. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιο μάθημα από εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπένιον. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς στη Ρωσία και η Ολλανδική ομάδα πάει εκεί και εντάξει, το καλύτερο. Στην Αφρική, στην ε, Ουγκάντα, πριν από ένα μήνα εγκρίθηκαν τα νομοσχέδια για τους ΛΟΑΔΜΟ. Εγώ μίλησα με ακτιβιστές από εκεί που είναι πραγματικά από τους σπουδάτερους ανθρώπους που γνωρίζω και ζητούν απελπισμένα τη βοήθειά μας. Στην Ιγερία, όπου η Γερουσία ενέκρινε νόμο που ποινικοποιεί όλες τις δραστηριότητε ΛΟΑΔΜΟ. Πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Ακόμα και στην Ινδία, όπου το νότατο δικαστήριο ποινικοποίησε και πάλι την ομοφιλοφιλία. Νομίζω ότι οι εξελίξεις σαν και αυτές που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ινδία πάνε χέρι το χέρι με περισσότερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, όχι αυτόματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει να κάνει πολλά ακόμα για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ. Εμείς έχουμε την ισότητα στις συνθήκη μας. Έχουμε και χρέος να βοηθήσουμε όλους τους καταπιεσμένους. Και δεν είναι η έννοια αγορά, η οικονομία αυτό για το οποίο πρέπει να απενεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τις αξίες της και αυτές πρέπει να μας καθοδηγούν σε σχέσεις που έχουμε με άλλες χώρες όπως με την Ουγκάντα, την Ιγυρία, την Ινδία και σίγουρα με τη Ρωσία. Ζητάω λοιπόν από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να αποποινικοποιηθεί η ομοφιλοφιλία σε ολόκληρο τον κόσμο και να υπάρχουν ίσα δικαιώματα για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κορνέλισεν. Ο επόμενος ένα λεπτό ο κύριος Κλάις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι πατέρας δύο μικρών παιδιών και ακούω τη δουλειά που κάνουν οι διάφοροι ΛΟΑΔΜΑ που καταπολεμούν την ε, ομοφοβία. Ένας όρος που δεν μ' αρέσει. Είναι ντροπή. Άνθρωποι το 2014 να ποινικοποιούνται και να διώκονται για τέτοιους λόγους. Σε 70 χώρε θεωρείται έγκλημα η μορφιλοφιλία. Σε αφρικανικές κυρίως χώρες, οι χώρες του Ισλάμ, που θεωρούν ότι μόνοι έχουν την αλήθεια. Διάφοροι συνάδελφοι εδώ που θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί πρέπει να αντί να ρίχνουν εκνοκοδίλια δάκρυα να δουλέψουν για να πάψει παραβίαση αυτή. Είναι το τελευταίο βήμα προκειμένου να καταλήξουμε σε μια σωστή λύση για το πρόβλημα. Για ένα λεπτό κύριε Γκέργκερντε Ούντμερκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε 78 χώρες απαγορεύονται οι σεξουαλικές πράξεις μεταξύ συνενούντων ε, ενηλίκων. Σε 7 από αυτές τις χώρες είναι κολάσιμες με την ποινή του θανάτου. Υπάρχει και διάκριση εναντίον των ε, θυμάτων βίας σε όλα στις χώρες αυτές όπου υπάρχουν κατασταλτικοί νόμοι στις ε, χώρες και νέοι νόμοι αυτού του είδους έχουν εγκριθεί στην Ιγυρία, στην Ινδία και στην Ουγγάντα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ενιαία και απαράγραπτα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει προστασία της σεξουαλικής ταυτότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζητά τον χωρί όρια σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να ενισχύσει την μη διάκριση κατά τον ΛΟΑΔΜ. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτά τα δικαιώματα όταν γίνονται σχέσεις και συμφωνίες με χώρες που έχουν αυτά τα προβλήματα. Κύριος Κάσμαν λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αυξανόμενη ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜΑ ε, είναι πραγματικά φρικτή. Στις τελευταίες 24 ώρες πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους απλώς και μόνο επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. Άλλοι φυλακίστηκαν στην Ιγυρία γιατί ακριβώς και μόνο είναι μόνο ε, ΛΟΑΔΜΑ. Ε, ο κύριος ε, Μπένιον αναφέρεται στην συνθήκη του, αναφέρθηκε στη συνθήκη του Κοτονού, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καθόλου διάλογος όσον αφορά τα δικαιώματα του ΛΟΑΔΜΑ. Θα πρέπει, είχαμε αναφέρει μία ρήτρα ήδη από το 1996 ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία εάν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ όμως έχουμε πραγματικά κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα που ξεκινάει η τρίτη ε, αναθεώρηση ε, θα πρέπει να εισακουστεί ε, η απέτησή μας να ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία αυτά στην αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και στη σχέση μας με τις χώρες ΑΚΕ. Διακόπτει ο μικρόφωνο στον Πρόεδρο του κ. Κωσούνα. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στη διαδικασία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ιερή η ανθρώπινη ζωή και δεν μπορεί να παραβιάζεται. Όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να εμποδίζουν να υπάρχει διάκριση μεταξύ ορισμένων ομάδων ανθρώπων και να υπάρχει παρότριση προς τη βία και το μίσος επί τη βάση σεξουαλικής προτίμησης. Γνωρίζουμε ότι σε πάρα πολλέ χώρε βέβαια οι ομοφιλοφιλικές σχέσει θεωρούνται έγκλημα, πολλέ φορέ ακόμα και με θανατική ποινή. Στην Ουγγάντα, στην Ιγυρία έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα οι νομοθεσίε και βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται στη Ρωσία όπου απαγορεύεται οτιδήποτε που αποτελεί προπαγάνδα υπέρ της ομοφιλοφιλίας χωρίς κανείς να καθοριστεί ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή <clears throat> η τάση για να δημιουργηθεί φόβος μεταξύ του πληθυσμού και να υπονομευθούν τα δικαιώματα των πολιτών. Βλέπουμε όλο και περισσότερες δρα... ενέργειες δράσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική ταυτότητα. Θα πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο ανεξάρτητα από την ε, προσανατολισμό μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχει τελειώσει η διαδικασία Κατσδιάη και δίνω το λόγο στον Επίτροπο Κέλλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την παραβίαση δικαιωμάτων ε, λεσβιών, μοφιλόφιλων, αφιλόφιλων, διφιλικών και μεσοφιλικών. Όπως δείχνουν τα πρόσφατα παραδείγματα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, ταυτότητα, τη σεξουαλική ταυτότητα κτλ. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται σαν άλοθη για παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ΛΟΑΔΜΑ εξακολουθούν να αποτελούν θύματα διώξεων και διακρίσεων σε πολλά μέρη του κόσμου. Σε 80 χώρες του κόσμου ποινικοποιούνται οι σχέσεις μεταξύ του δύο φύλου Έχουμε και παραδείγματα και πιο πρόσφατα με νομοθεσία που έχει εγκριθεί στην Ιγυρία για παράδειγμα για αυτό το θέμα. Πρόσφατα επίση έχουμε ακούσει και παπανικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο φίλων και αλλού. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά είναι ασύμβατα με την νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω και εμεί πρέπει να δράσουμε. Ακριβώς Γι' αυτό έχει αρχίσει και πάλι η συζήτηση για τους περιορισμούς αυτούς που είναι απαράδεκτοι και όπως ξέρετε, το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου του 2013 έκρινε κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΟ. είναι κάτι που βρίσκεται στην καρδιά των πολιτικών μας και για το λόγο αυτό έχουμε διάφορα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πατός ε, εκπρόσωπος έχει κάνει δηλώσεις σχετικά όπως τον Ιούνιο για παράδειγμα όπου εγκρίθηκε ο νόμος κατά της προπαγάνδας στη Ρωσία ή μετά από την δράση της Ινδίας επ' αυτού και τον Δεκέμβριο μάλιστα σχετικά με την ομοθεσία της Ουγκάντα και ακόμα και χτες όταν υπογράφτηκε κάτι σχετικό και στην Νιγηρία που περιορίζει τα δικαιώματα αυτά. Είναι και θέματα επίσης που αναφέρονται στους διαλόγους που έχουμε με τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα τη Ρωσία και την Νιγηρία, για αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε και να στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών μέσω των εργαλείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν οι προτάσεις λοιπόν για στήριξη των ατόμων αυτών και οικονομική ήδη από τον Αύγουστο του 2013 για 5 εκατομμύρια και θα συνεχιστεί και το 2014. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πρόθεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ώστε να μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν οι άνθρωποι τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να στηρίζουμε. Δεν μπορεί να σιωπούμε Όσον αφορά την άρση του άρθρου 96 στη συνθήκη Κοτονού, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να δούμε πρώτα όλες τις άλλες δυνατότητες που έχουμε για να επηρεάσουμε τις εξελίξεις πριν φτάσουμε σε αυτήν την ε, τελευταία από τις λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Κάλλας. Περνάμε τώρα μάλλον έχουμε έξι ψηφίσματα για την λήξη της συζήτησης. Τώρα θα λάβει χώρα αμέσως η ψηφοφορία των ψηφισμάτων. Ερχόμαστε πρώτα στην ψηφοφορία σε σχέση με την κατάσταση στην Καμπότζη και το Λάος. Έχουμε το κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων, τροπολογία